άρθρου του αρμόδιου του, κοινοβουλίου, του, του εάν μια πολιτική ομάδα ή 40 βουλευτές δεν, θέσουν, δεν γίνουν εγκύρηση, το κείμενο αυτό θα θεωρηθεί ότι έχει εγκριθεί. Θα προσαρτηθεί το κείμενο στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Έχουμε τώρα μία αίτηση για διαδικαστική ε, παρέμβαση από τον κύριο Γλέζο. Παρακαλώ κύριε Γλέζο. Συνάδελφοι, 1100 παιδικοί σταθμοί με 5.500 παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύουν να μην λειτουργήσουν από έλλειψη εφοδίων. Και, και ενώ αυτή είναι η κατάσταση και ενώ έπρεπε να ασχοληθεί η Κομισιόν ειδικά με αυτό το θέμα και με άλλα παρόμοια που ταλανίζουν τους λαούς της Ευρώπης, ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ ως υπερεξουσιαστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχείρησε με απαράδεκτες αντιδεοντολογικές και αντιδημοκρατικές επεμβάσεις να κατευθύνει το ελληνικό κοινοβούλιο. Με ποιο δικαίωμα επιχειρεί να βιάσει αν όχι με που επειδή έχει τώρα ε, βοηθούς τους συγκυβερνήτες, τον πληροφορώ ότι δεν θα μπορέσει να το κάνει μεθαύριο που στην εξουσία θα είναι ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Κύριε Γλέζο, λέει ο πρόεδρος. Αγαπητέ συνάδελφοι. Είναι. Είναι χρήσιμο το γεγονός ότι θέλετε να κάνετε αυτή την παρέμβαση, αλλά αυτό το περιεχόμενο της ε, παρέμβασής σας θα πρέπει να είναι διαδικουστικού χαρακτήρα και όχι μια πολιτική παρέμβαση. Είναι η κλασική περίπτωση χρήσης των ε, αγορεύσεων ενός λεπτού. Κύριε Γλέζο, αν θέλετε να λάβετε το λόγο για ένα τέτοιο θέμα, σας παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία των ομιλιών ενός λεπτού. Ευχαριστώ πολύ, λέω ο Εάν δεν υπάρχει περαιτέρω παρέμβαση για πραγματικά διαδικαστικό θέμα, κύριε Λάμπερτς, για διαδικαστικό θέλετε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Εξ ονόματος της ομάδας μου ζητώ να μπει στην ημερήσια διάταξη της τωρινής Ολομέλειας συζήτηση και ψήφισμα για το πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν. Ούτε και αυτό για την ημερήσια διάταξη. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ημερήσια διάταξη της εβδομάδας αυτής. Κοιτάξτε. Καλά, καλά το προσπαθήσατε, αλλά και εγώ ήμουν πρόεδρος πολιτικής επιτροπής, ξέρω τα παιχνίδια, αλλά πρέπει να ακολουθούμε τη σειρά τη ημέρας τη διάταξη. Ερχόμαστε στο, στο σημείο.